να κάνω. Ο κ. Ζανλούκα Μπονάνο, μέλος του Κοινοβουλίου, υπέβαλε έτοιμα στον Πρόεδρο για υπεράσπιση της ασυλίας του στα πλαίσια ποινικών διώξεων από το δικαστήριο του Μπολτζάνο. Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό, το αίτημά του παρεπέμφθη στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων